Ε, είναι διαθέσιμα και θέλω να σα ρωτήσω αν υπάρχουν αντιρρήσει ή παρατηρήσει για τα πρακτικά. Αν όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει